good afternoon. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Έχω τη χαρά να αντικαθιστώ για σήμερα τον Κλοντ Μωράης, ο οποίος είχε κάποιες απρόβλεπτες υποχρεώσεις. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να γίνει εξή ε, αλλαγή στην μέση διαταξή, να σα είναι την εξή αλλαγή. Παρουσίαση τη Επιτροπή για τη νέα συνεροφυλακή και ακτοφυλακή με εισηγήτρια την κυρία Μετσόλα, σημείο 5, θα ξεκινήσει στι 3 αντί για τι 4.30, δηλαδή τώρα. Και στο σημείο 8, η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότηση προστασία ατόμων ε, που καταγγέλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 18 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται. Άλλο σημείο. Σας παρακαλώ, σημειώστε ότι η διερμηνία θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες ε, πλην κροατικών, δανικών και γελικών. Και μια άλλη παρατήρηση. Ε, διορισμός εισηγητών για τις συστάσεις. Μαρία Γκραπίνη, εισηγήτρια για την γομοδότηση της έκθεσης ΑΦΚΟ, για την έκθεση ε, εφαρμογής των νομικών διατάξεων και τη κοινή δήλωση που εξασφαλίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τους αποκεντρωμένου οργανισμού. Εγκρίνει τη σύσταση αυτή Τη εισηγήτρια η Επιτροπή μα ωραία. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία σήμερα στι 5 και 4. Παρακαλώ, φροντίστε να είστε εδώ και να έχετε και τι κάρτε σα για να ψηφίσετε. Επόμενο σημείο, βασικό σημείο, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Πριν από δύο χρόνια, οι δύο συνομοθέτε έφτασαν σε συμφωνία για τη δημιουργία νέα συνεροφυλακή και ακτοφυλακή. Και αυτό στο απόγειο τη ε, μεταναστευτική κρίση το 2015. Έρχονται κατάσταση στα εξωτερικά μα σύνορα άλλαξε σημαντικά. Ωστόσο, η Μεσόγειος παραμένει ένα μέρος όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ε, διακινδυνεύουν τη ζωή τους ετησίως. Περαιτέρω βήματα χρειάζονται ως μέρος της ε, σφαιρικής προσέγγισης για να διαχειριστούμε τα σύνορα. Ε, την περασμένη εβδομάδα οι Ευρωπαϊκοί Σύνοροφυλακοί και Ακτοφυλακοί γιόρτασαν ε, τα γενέθλιά τους δύο ετών. Κατά τα δύο αυτά χρόνια ο οργανισμός αυτός έχει αναλάβει πλήρως και έχει περίσπερα στην εντολή του. Το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμά του 30 Μαΐου 2018 για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν εξέφρασε τις ανησυχίες τους ό,τι αφορά την εφαρμογή της εντολής. Η ανησυχία αυτή έχει να κάνει περισσότερο με τις ε, πλημελείς δεσμεύσεις των κρατών μελών που δεν συνεισφέρουν με αρκετούς ανθρώπινους πόρους και τεχνικό εξοπλισμό για τις κοινέ επιχειρήσεις και την ταχεία αντίδραση στη σχετική συγκέντρωση δυνάμεων για ταχεία απόκριση. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να ενισχυθεί ο ρόλο του οργανισμού κατά τη διάρκεια τη τρέχουσα θητεία του. Το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να ε, ενισχύσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση για την σενεροφυλακή και την ακτοφυλακή. Ε, σήμερα η Επιτροπή είναι εδώ για να σχολιάσει την πρόταση και να απαντήσει στι ερωτήσει μα. Ο, ρόλος, ο λόγο στον κύριο Ντεκόιστερ από την Επιτροπή για 10 λεπτά. Did I pronounce it correctly? Μήπως δεν το πρόφερα σωστά. Περίπου. Problems with my name sometimes, so people are... Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, good... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Τιμή και χαρά να σας παρουσιάσω εδώ σήμερα την άποψη της ε, πρότασης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Σεπτεμβρίου. Μου δώσατε τα 10 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι αρχικά τα, μέρη της, τα μέλη της ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να πάρουν το λόγο για να κάνουν ερωτήσει σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Φυλακή και Εκτοφυλακή. Αλλά τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για μένα προσωπικά και ύστερα. Και μόνο το κεφάλαιο να σας διαβάσω. Τους τίτλους των κεφαλαίων της πρότασης ε, θα μου χρειάζονταν 10 λεπτά. Παρ' όλα αυτά να κάνω ό,τι μπορώ και είμαι βεβαίως ότι πρόκειται μόνο για μια πρώτη παρουσίαση, μια πρώτη έτσι, επαφή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ερωτήσεις που έχετε σε ό,τι αφορά το πολιτικό συγκείμενο σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς το εξής. Να αναφερθώ στην ομιλία του Πρόεδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, όπου στο Κοινοβούλιο ανέφερε ότι πρόκειται να υπάρξει ένα νέο πακέτο μετανάστευσης, το οποίο θα ενέκρινε στις 12 Σεπτεμβρίου το Σώμα των Επιτρόπων, που θα κάλυπτε πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τις νόμιμες οδούς εισχώρησε στην Ένωση και τόνισε ε, ότι μόνο συλλογική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σημειώσει διαφορά επιτόπου. Μας υπενθύμισε επίσης ότι το πακέτο αυτό μεταφράζει το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πουδουπού. Μία προτάση που ενεκριθεί στις 2 Μαΐου για μια ενισχυμένη συνοριοφυλακή και αυτοφυλακή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 10.000 μόνιμους συνοριοφύλακες. Πρόεδρο. αυτά λέει η πρόταση. Αυτό και είναι και το βασικό στοιχείο της πρότασης του πακέτου του Σεπτεμβρίου. Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χρησιμοποίησαμε EBCG 2.0 ως τίτλο εργασίας. Το EBCG 1,0 είχε εγκριθεί το 2016 και έτσι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ευρώπη μοιάζει με παραγωγό iPhone. Κάθε δύο χρόνια βγάζει και μια καινούργια εκδοχή. Το πιο προφανές λοιπόν ερώτημα είναι το εξή. Αν το EBCG 1.0 εγκρίθηκε από τις νομοθέτες το 2016, γιατί σήμερα ήδη προκύπτει η δεύτερη ερώτηση για το 2.0. Και ίσως, Πρόεδρε, να είμαι σύντομος σε ό,τι αφορά το πιο σημαντικό στοιχείο της πρότασης. Αυτό το μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων και άλλων μελών προσωπικού. Η αναγκη υποβολή πρόταση καταρχά, ε, καταρχάς, γιατί υπάρχουν 5-6 λόγοι, αλλά ο πρώτος, λόγος, ο πρώτο και καλύτερο είναι η αποτυχία εφαρμογή και υλοποίησης του EBCG 1.0, του σχετικού κανονισμού. Μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις τη ε, της ε, πρότασης είναι να εξασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία θα έχει στη διάθεσή της επαρκείς τεχνικούς πόρους, για να εκτελεί τις δράσεις που απαιτούνται για να υποβοηθηθούν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την προστασία των τμήματων που τους αναλογούν στα εξωτερικά σύνορα. Το είπατε και εσείς, Πρόεδρα, εισαγωγικά. Κατά τα δύο χρόνια που έχουμε πίσω μας, η υπηρεσία αντιμετώπισε μεγάλα κενά και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις τεχνικές προδιαγραφέ ε, για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά τη. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Υπήρξε μια πολύ σημαντική βελτίωση στο κείμενο. Τότε που δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα 1500 συνοριοφυλάκων για ταχύα αντίδραση. Αυτό μάλιστα ήταν ένα στοιχείο. Δεν εφαρμοστήκε όμως από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ασυνοριαφυλακής και Ακτοφυλακής της πρώτης έκδοσης. Γιατί? Γιατί πρόκειται μόνο για ταχείες αντιδράσεις, όχι για τις κανονικές ενέργειες και δράσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Άρα υπήρξαν κοινέ δράσεις και σωστές υποδομές, αλλά αυτό έπρεπε να προέλθει από την εθελούσια συμμετοχή των κρατών μελών. Αυτό προφανώς δεν αρκεί και είναι απαράδεκτο αν θέλουμε να προετοιμάσουμε μελλοντικές καταστάσεις. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αυτή την ιδέα ενός μόνιμου σώματος δεκαχιλιάδων φυλακών. Γιατί 10.000, να σας το πω. Στο σύστημα περιλαμβάνονται 7.000 μέλη προσωπικού από τα κράτη-μέλη που έχουν καταχωριστεί. Υπάρχει και η ομάδα ταχύς αντιδρασής 1.500 και άλλη μια ομάδα με 600-700 εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Αν ε, συνυπολογίσουμε και αυτά που είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι χρειαζόμαστε μηχανισμούς και μέσα που θα είναι αποτελεσματικά για την διαχείριση της μετανάστευσης. Δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία μόνο της ε, υπηρεσίας στις κοινέ δράσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι θα χρειαστούμε στο μέλλον και πιο πολλούς ανθρώπινους πόρους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν να συνεισφέρουν, να συμβάλλουν σε αυτό το μόνιμο σώμα. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά τι σημαίνει Φτάνει πια αυτό το θελούσιο σύστημα. Το σύστημα θελούσια συνεισφορά και συμβολή. Και πέραν τούτου έχουμε και άλλη μια σημαντική καινοτομία. Ότι το ίδιο το προσωπικό της Υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να καταστεί μέλος της ομάδας που θα αναπτυχθεί επιτόπου από την υπηρεσία. Θα είναι Ευρωπαίοι δηλαδή οι υπάλληλοι αυτοί που θα εκτελούν τις ε, επιχειρήσεις ε, επιστροφής ε, και φύλαξη των συνόρων. Είναι σημαντικό αυτό το καινοτομικό στοιχείο και θα είναι και το σημείο εφετηρίας για όλες τις μελλοντικές δράσεις. Αυτέ οι δυνατότητε λοιπόν θα είναι στη διάθεση τη υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και μία δεύτερη κατηγορία. Άτομα τα οποία θα είναι αποσπασμένα από τα κρατημέλη για μεγάλη διάρκεια. Και αυτοί θα είναι στη διάθεση τη υπηρεσία και έχουμε και μια τρίτη κατηγορία ατόμων, εμπειρογνώμων από τα κράτη-μέλη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινέ δράσει για πιο βραχαία χρονικά διαστήματα, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες και στο παράδειγμα εξηγείται πώς θα εξελιχθεί η σύνθεση αυτή με την πάροδο του χρόνου σε ό,τι αφορά το μόνιμο αυτό σώμα γιατί δεν ξεκινάμε με 7.000 άτομα νέο προσωπικό. Αυτό είναι αδύνατον άλλωστε. Πού να τους βρούμε μέχρι το 2020 για να τους ε, προσλάβουμε, γιατί το 2020 θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσταθεί αυτό το μόνιμο σώμα. Ένα σημείο να τονίσω. Υπάρχει μια κάποια παρανόηση για αυτή τη νέα πρώτη κατηγορία, το προσωπικό της υπηρεσίας αυτόνομο δικαίωμα για να δρουν στην επικράτεια των κρατών μελών. Αυτό που είναι καινούριο όμω είναι το εξή, ότι το προσωπικό τη υπηρεσία στο μέλλον θα είναι σε θέση να είναι τμήμα των ομάδων που ενεργούν επί τόπου. Δεν μπορούν όμω να μπουν στο κράτος μέλο, από του καπνίσει και να κάνουν ό,τι θέλουν σε ό,τι αφορά την επιστροφή, τον έλεγχο των συνόρων και το καθεξής. Όχι, προφανώ. Θα είναι μέλη τη ομάδα και θα είναι επίση όρις με τους εμπειρογνώμονες που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη-μέλη. Και πάλι, κάτι άλλο που θέλω να το τονίσω, γιατί υπάρχει μεγάλη παρανόηση στο σημείο αυτό. Το σύστημα αυτό δεν επηρεάζει το σύστημα κοινών ευθυνών, την αρχή της κοινής ευθύνη για τα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη σε πρώτη μοίρα για τη φύλαξη του, των συνόρων που τους αναλογούν, αυτό που εξασφαλίζεται είναι όταν θα χρειαστεί ενίσχυση από την υπηρεσία να έχει την ικανότητα να παρέχει υποστήριξη, αλλά οι ομάδε δεν μπορούν, επαναλαμβάνω, να μεταβούν στα κρατη και να δρουν αντί των μελών. Οι δράσει πάντα θα προαπαιτούν την αποδοχή και συνεργασία του εκάστοτε κράτου μέλου. Άρα αυτή ήταν η αποτυχία τη Ευρωπαϊκή Ιδρυνοφυλακή και και αυτό ήταν και ο πρώτο λόγο που μα οδήγησε στην ε, δημιουργία τη νέα αυτή μορφή. Να προχωρήσω γρήγορα και στα υπόλοιπα. Άλλη μια σημαντική καινοτομία, όχι τόσο επί της ουσίας, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συνόρων πλέον έχει ενσωματωθεί μετά από την ε, εξέταση του κανονισμού Eurosal μέσα στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία Φυλακή και Εθοφυλακή ήταν ε, ένας στάνταρ κανονισμός που παίζει σημαντικό ρόλο για την ε, παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και περιλαμβάνει και ένα μηχανισμό ανταπόκρισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κανονισμός θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη το 2016, αλλά λόγω της έγκρισης της πρώτης Ευρωπαϊκής Συνορία Φυλακής και Εκτοφυλακής αναβλήθηκε, αλλά συμπεριλεύτηκε και στο πακέτο του Σεπτεμβρίου αυτή η αναθεώρηση. Και υπογραμμίζει και τις αλλαγές που έγιναν στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Φυλακή και Καταφυλακή. Όπως θα δείτε δε, υπάρχουν και επαφέ σε ό,τι αφορά Αυτό που αναπτύξαμε είναι ο αντίκτυπο του κ. Eurosurs, ό,τι αφορά για παράδειγμα τον προγραμματισμό των ικανοτήτων, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και το καθεξή. Άρα, δεν μεταφέρουμε απλά αυτού ή τον αναγωνισμό σε έναν άλλον. Όχι, θέλουμε να υπάρχει πλήρη συνοχή και αξιοποίηση των ικανοτήτων τη Ευρωπαϊκή Συνοριαφυλακή και Εκτοφυλακή. Ένα τρίτο λόγο για την υποβολή τη πρόταση αυτή είναι ότι στον τομέα των επιστροφών δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Και όπως ξέρετε, η σωστή πολιτική επιστροφών είναι ένα βασικό στοιχείο, αναπόσπαστο θα έλεγα, της σωστής μεταναστευτικής πολιτικής. Άρα, παρά το γεγονό ότι τονίστηκε και ενσωματώθηκε ο ρόλος της Ρεφλέγης και το φυλακή και στην πρώτη έκδοχη, θα πρέπει να τον ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω. Σε διάφορα κεφάλαια λοιπόν θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν τέτοιες ε, πρόσθηκες για την επιστροφή σε ό,τι αφορά την εντολή της υπηρεσίας. Ένα άλλο στοιχείο σε ό,τι αφορά τις εξεκλήξεις. Το θέμα που είναι πολύ βασική ε, και θεμελιωδού σημασία για την ευρωπαϊκή διαχείριση της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απομονωμένοι. Χρειάζεται συνεργασία με τρίτε χώρε. Στην πρώτη Ευρωπαϊκή Συνεργασία Φλαϊκή υπήρχαν διατάξει για τη συνεργασία με άλλε γειτονικέ χώρε με δυνατότητα ανάπτυξη επιχειρήσεων στην επικράτεια τρίτων χωρών. Αλλά φυσικά υπό την αίρεση τη συμφωνία. Πέντε τέτοιε συμφωνίε έχουν συναυθεί με χώρε Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα πλέον στην πρότασή μα Υπάρχει η προδιαγραφή για γειτονικέ τρίτε χώρε ε, η υπηρεσία. Μάλλον ε, δεν υπάρχει πλέον αυτή η απέτηση να είναι γειτονική αυτή η τρίτη χώρα. Είναι πολύ ευαίσθητο σημείο αυτό, το ξέρω. Και η δυνατότητα συνεργασία με τρίτε χώρε στον τομέα των επιστροφών αναπτύσσεται περαιτέρω στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήταν και στην πρώτη πρόταση, δεν είχε συμφωνήσει ο συνομοθέτη, αλλά από ό,τι βλέπετε υπάρχουν καλοί λόγοι να ξανανοίξει αυτή η συζήτηση για κάποια τα θέματα αυτά. Τα χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. Υπάρχει επίσης και θα περιοριστώ στο σημείο αυτό σε μία πρόταση. Υπάρχει σήμερα και το ΦΑΝΤΟ, ένα ευρωπαϊκό σύστημα απεικόνησης για την, ε, τα γενικά έγγραφα και πάλι βασιζόμαστε σε μια κοινή δράση από τη δεκαετία του 90 μάλιστα θα πρέπει να περάσει από τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορεί δηλαδή να διαχειρίσετε το, το Συμβούλιο την ατζέντα αυτή και προτείνουμε επίση και η Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Συνοριαφυλακή και Φυλακής να καταστεί υπεύθυνη και αρμόδια για την διαχείριση του συστήματο αυτός. Τελευταίο λόγο για τι αλλαγέ που προτείνουμε που φυσικά επηρεάζουν πολλές διατάξεις σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, τον πρώτο, την ευρωπαϊκή ιστοριοφυλακή και Εκθοφυλακή και με σημαντικό αντικτύπο μάλιστα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε και την διαχείριση, την διακυβέρνηση της υπηρεσίας, γιατί κάποιοι λένε ότι προτείνουμε ένα τέρας, πολλά χρήματα, πολλές ευθύνες, πολλές αρμοδιότητες, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο και να δοθεί πολιτική καθοδήγηση στην υπηρεσία για όλα αυτά τα θέματα. Και στο θέμα λοιπόν των διατάξεων διαχείρισης έχουμε επιφέρει σημαντικέ αλλαγέ. Πρόεδρε, αυτά. Πολύ, πολύ, πολύ συνοπτικά. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους προτείναμε αυτά που προτείναμε. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο που κατανόησε με σαφήνεια πόσο κατεπίγουσα είναι αυτή η πρόταση και που όρισε στο συντομότερο χρονικό διάστημα την εισηγήτρια. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σα πω ότι είμαστε απόλυτα διαθετημένοι να κάνουμε όσο πιο πολλέ ε, και όσε συναντήσει χρειαστούν για να απαντήσουμε σε όλε τι ερωτήσει που ενδεχομένω να έχουν οι βουλευτέ. Πλήρη διαθεσιμότητα και προθυμία συνεργασία από πλευρά μα. Θα διευκολύνουμε και λυπάμαι που κλείνω με ένα τόσο βαρετό σχόλιο. Πολλά στοιχεία είναι καινούργια στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τον παλιό κανονισμό, αλλά και υπάρχουν και πολλές διτάξεις που δεν τις αγγίξαμε καθόλου. Και φυσικά, όταν διαβάζετε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να μην είναι σαφές ε, τι υπάγεται πού, σε ποια κατηγορία. Άρα τις επόμενες ημέρες θα σας δώσουμε ένα εγγράφο με παρακολούθηση αλλαγών δεν έχει νομική υπόσταση. Θα σας ε, επιτρέψει όμως να κατανοήσετε τι ισχύει ήδη, τι ισχύει από τον πρώτο κανονισμό και τι άλλαξε και δούλεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά, Πρόεδρε, ελπίζω να κατάφερα να σας δώσω μια ιδέα για τον κανονισμό, για την πρότασή μας και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν ε, φοβερά ε, κατατοπιστική η ανάλυση σας. Ξεπεράσατε τα 10 λεπτά. Αλλά ήταν απαραίτητο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα. Για την ώρα δεν ζητά κανείς το λόγο. Μάλλον όχι, η κυρία Μετσόλα, ο κύριος Νίντερ Δεν βλέπω ποια άλλη θέλουν το λόγο για την ώρα. Κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την εξαιρετική παρουσίαση. Νομίζω, αν δούμε πώς εξελίχθηκε η Frontex, έχει κάνει φοβερή πρόοδο, έχει αναπτυχθεί και τώρα αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμω να εξυγχρονίζουμε τη Frontex και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών τη. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα όλα αυτά να έχουν γίνει καθαρά και εξάστερα πριν τις εκλογές του Μαΐου και να είμαστε ε, έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι παρόλο που το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλαγέ πρέπει να γίνουν γρήγορα για να μπορέσει ο οργανισμός να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά του και να προστατεύει τα εξωτερικά μας σύνορα. Θα πρέπει με μια γρήγορη διαδικασία ε, ο οργανισμός να αναλάβει τις επιπλέον αρμοδιότητες και να λειτουργεί πλήρως ως το 2020. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να τη χάσουμε, διότι τελικά κανείς δεν θέλει έναν σούπερ οργανισμό που δεν θα λειτουργεί όμως. Θέλουμε να μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στα επιπλέον που ανέλαβε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση μπορούμε να χτίσουμε σε αυτά που ήδη είχαμε στα χέρια μας και σε αυτά που προτάθηκαν. Θα βελτιώσουμε το σύστημα και θέλουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσής μας. Ε, η βελτίωση τη αποτελεσματικότητα είναι σημαντικό. Όμω πρέπει να σεβαστούμε και τι αρμοδιότητε και ευθύνε των κρατών μελών. Δεν θα προτείνουμε καμία μετατόπιση στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο ρόλο και οι υποχρεώσει των κρατών μελών βάσει τη εθνική νομοθεσία, όπω με τη Σύμβαση για τον νόμο τη θάλασσα ή για την ασφάλεια τη ζωή στη θάλασσα ή για τη θαλάσσια διάσωση, τη διάσωση και την ε, προστασία στη θάλασσα δεν έχουν αλλάξει. Είναι φιλόδοξη η πρόταση να αυξηθεί το προσωπικό του οργανισμού. Γιατί όμως θα πρέπει να βασιστεί στα κράτη-μέλη ε, ο οργανισμός για να έχει ε, επάνδρωση εκεί που χρειάζεται. Εάν κοιτάξουμε τους αριθμούς για να είμαστε βέβαιοι ότι έχει 10.000 ε, μόνιμους υπαλλήλου, θα πρέπει να δούμε ότι ο αριθμός είναι ρεαλιστικός για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του οργανισμού. Δεν μιλάμε για λειτουργικούς που θα είναι διαρκώς ε, σε επιχειρήσεις την ίδια στιγμή. Πρέπει να δούμε και τη σύνθεση του μόνιμου προσωπικού. Θα πρέπει να έχουμε ε, αποσπασμένους για μικρότερα και μεγαλύτερα διαστήματα και να σκεφτούμε και τι πόρους θα χρειαστούν για να αντικατασταθούν στις χώρες τους. Ή μήπως οι πόροι θα πρέπει πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, για τον οργανισμό, να εκπαιδεύσει τους μόνιμους υπαλλήλου του και ε, τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν αυτούς που ήδη έχουν και είναι έμπειροι. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Επίσης, το θέμα δεν είναι πια ποιους υπαλλήλους τα κράτη-μέλη θα στείλουν αμέσως, αλλά και θα υπάρχει ο τεχνικός εξοπλισμός σε αυτό που είναι αυστηρός απαραίτητο για να ξεκινούν αμέσως οι αποστολές χωρίς καμία καθυστέρηση. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε περισσότερα κονδύλια για τους οργανισμούς, επιπλέον υποχρεώσεις και ευθύνε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ε, μεγαλύτερο και ενισχυμένο προπολογισμό. Αυτό που με εκπλήσει είναι που ο οργανισμός ήδη μπορεί να αποφασίσει μπορέσει να τον τεχνικό του εξοπλισμό. Αυτό θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει από το 2011, όμως ε, δεν μπορούσε γιατί δεν είχε πάρει τους δημοσιονομικούς πόρους που χρειαζόταν. Ένα άλλο στοιχείο τη πρόταση αυτή είναι η επικέντρωση στι επιστροφέ. Θα πρέπει οι αριθμοί των επιστροφών να αυξηθούν. Η προστασία πρέπει να χορηγείται σε όποιον την ε, χρειάζεται, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να επιστρέφουμε όσου δεν ε, χρήζουν τέτοιε προστασίε αμέσω και γρήγορα. Θα πρέπει ο οργανισμό να αναλάβει εδώ το ρόλο του για να γίνεται αυτό σωστά. Αν δω την Μάλτα, που είναι μικρή χώρα και δεν έχει διπλωματική εκπροσώπηση σε όλες τις χώρες προέλευσης όπου πρέπει να επιστρέψουν οι πρόσφυγες, ε, Εκεί είναι που ένας τέτοιο οργανισμός μπορεί να βοηθήσει τη Μάλτα, το, τη χώρα μου όπως και τόσες άλλες, να ετοιμάσει τα έγγραφα αυτών των ανθρώπων που πρέπει να επιστρέψουν. Όσων δεν εκπληρώνουν τις προποθέσει για τη διαμονή και την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι τα μόνα που θα λαμβάνουν την τελική απόφαση. Αυτό όμω πρέπει να κάνει ο οργανισμό είναι να διευκολύνει τη διαδικασία για να μπορούν να ληφθούν τέτοιε αποφάσει. Όλες αυτές οι πρόσθετες αρμοδιότητες πρέπει να αναλυθούν... σε πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει εδώ να επιταχθεί κάποια συμφωνία. Ο οργανισμός έδειξε ότι είναι μία από τις προτεραιότητές του, τον έχουμε ενισχύσει ε, στην υπηρεσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ισκα Κέλλερ και εγώ ίδια πιέσαμε στο οργανισμό να εφαρμόσει ένα μηχανισμό προσφυγής, επίλυση διαφορών, που ήδη προβλεπόταν στην πρόταση τη Επιτροπής πριν από δύο χρόνια. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε να βεβαιωθούμε ότι ο οργανισμό και αποτελεσματικό θα είναι και θα σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι πάρα πολλά που μπορώ να πω για ένα τόσο ευρύ θέμα. Βλέπω που νεύεται, αλλά πολύ σύντομα μια-δυο ακόμα παρατηρήσει ε, και μετά θα ολοκληρώσω. Η συμπερίληψη του Eurosol στους ε, οργανισμούς αυτούς είναι σημαντικό να έχουν εθνικά κέντρα συντονισμού τα κρατημέλη για να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, είναι διαλειτουργικά τα συστήματα, ο οργανισμός να συνεργάζεται με τρίτες χώρες για να τη στηρίζει στη διαχείριση των σύνορων, την μετανάστευση και τις επιστροφές και τέλος πρέπει να βρούμε τρόπους για να γίνει ο οργανισμός ένας ελκυστικός χώρος εργασίας. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει ο οργανισμός για την πρόσληψη. Το σύστημα θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο για να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού και ταυτόχρονα βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση με, ε, σε σύγκριση με άλλους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η πρώτη συνάντηση σκιωδών. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους τους σκιώδεις από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για να υπάρχει ε, μια κατάλληλη επίλυση, ένα κατάλληλο πέρα στην όλη διαδικασία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε να μας τα παρουσιάσει αλλά και την ε, εισηγήτρια για την τόσο πλήρη παρουσίασή της να μην μπούμε στις λεπτομέρειες απλώς πρέπει να σας πω ότι 28 εκ του 16 Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συνεφώνησαν όσον αφορά την ακτοφυλακή και την οριοφυλακή όπως μας τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης είναι πάρα πολύ θετικό ότι όλα προχώρησαν και διεκπαιρέθηκαν γρήγορα. Έχουμε την Frontex και τώρα έχουμε τη νέα πρόταση μετά από δύο χρόνια ούτως ώστε να βαθμίσουμε την αντολή της Frontex. Ε, όλα αυτά αποτελούν μια ε, ερμηνεία πάρα πολύ κομψή. Έχουμε τώρα ε, την Frontex 2 μηδέν δεύτερη γενιά δηλαδή, ε, που δεν είναι iPhone. Ε, δεν είναι iPhone η Frontex, δεν θέλει δηλαδή την επικαιροποίηση που θέλει συνέχεια το iPhone. Τέλος πάντων, έχουμε τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου του Ζάλσμπουργκ και όλα αυτά χρειάζονται για τα κράτη-μέλη. Και δεν χρειάζονται και άλλες παραχωρήσεις και δεσμεύσεις. Άρα αλλάξαμε διάφορα πράγματα στη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια ε, ανάλογα με το τι ζήτησε και η Eurostat. Έχουμε τώρα την τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Ε, έχουμε και την λύση για τον τελείω νέο κανονισμό. Μα γιατί. Τότε γιατί το 2016 κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Έχει κάποιες παλιές ιδέες η Κομισιόν όσον αφορά κάποιες επιστροφές κάποιων πίσω στις χώρες τους. Ε, ε, οι συνομοθέτες πάνε όχι σε αυτό. είπαμε για 10.000 το είπε και η κυρία Μετσόλα ως προσωπικό αλλά από πού βγαίνει αυτό το νούμερο έχει γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων αλλά δεν το είχε γίνει για τον προηγούμενο οργανισμό. θα πρέπει να το συνηθίσουμε έχει διαβρεθεί εντολή από το 16 της Frontex και η ΆΣΟ επίσης λειτουργεί εκτός εντολής εδώ και κάποια χρόνια το μεταναστευτικό έχει ωφελεί στην υπηρεσία. Άραγε. Τέλο πάντων, έχω πολλέ επιφυλάξει αυτή την πρόταση και ιδίω για το πώ έγιναν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ο νέο κανονισμό πρόκειται να μα δώσει τίποτα έξτρα. Κάποια προσθέμενη αξία τέλο πάντων. Κύριε Δεπρέ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα. να συμπαθάτε τη σκιώδη εισηγητριά μας, την κυρία Ναταλή Γκρισμπέκ, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Και αν κατάλαβα καλά, δεν θα έρθει και στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών που θα λάβει χώρα αμέσω μετά. Και να σας πω εκ μέρους της τάξης πριν από 10 χρόνια, 6 το 7, είχαμε ένα πρόγραμμα, το λέγαμε Rabbit και του Rabbit ήμουν εγώ εισηγητή. Τι ήταν, ήταν το πώ τα κρατημέλια θα μπορέσουν να αποδεσμεύσουν κάποιους συνοριοφύλακε και να τους ε, αποσπάσουν εκεί σε μια τέτοια υπηρεσία όπως το συζητούμε. Δεν τους άρεσε αυτό πολύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα δε κράτη-μέλη ήταν 100% ε, κατά τα πράγματα έχουν ε, εξελιχθεί από τότε. Έχουμε όμως τέσσερα ερωτήματα σχετικά με αυτό. Τι καθεστώς διέπει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Τι γίνεται, τι, τι, τι καταστατικό έχουν. Έχουμε τις εθνικές υπηρεσίες, τρεις κατηγορίες. Πώς θα συγκατοικήσουν, πώς θα συνεπάρξουν τόσες υπηρεσίες που έχουν τόσο διαφορετική φύση και οι εθνικές υπηρεσίες ασχολούνται με τα σύνορα στις περισσότερες χώρες. Τι λέει η Επιτροπή. Αυτό το πρόγραμμα που τώρα χαράσετε θα ισχύσει και στο απότερο μέλλον. Ας το κοιτάξουμε το θέμα. όσο με τώρα τις επιστροφές, τους επαναπατρισμούς, αυτό που πραγματικά είναι νέο Ποιο είναι, μιλάτε για καινούριε αρμοδιότητες ή για κινητοποίηση επιπλέον προσωπικού, διεύρυνση αρμοδιοτήτων νέου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, μεταξύ 16 και 17 έχουμε μείωση των επιστροφών αυτών. Τώρα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ε, βέβαια θα πρέπει να θεωρηθεί θετικό ότι η συνεργασία περνά από τη συμφωνία με την εκάστοτε χώρα. Τι ισχύει κάτι τέτοιο με τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, περισσότεροι έρχονται από τον Νότο. Άρα εκεί είναι η πιο επιτακτικές ανάγκες. Προς αυτή την κατεύθυνση. Euh, τι, τι εννοείται για ένταξη της ρύθμισης στο καθεστώς της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ο ίδιος σκιώδης εισηγητής και δεν έχω μελετήσει την ουσία τη πρόταση. Ο πρόεδρο. Έχω μια σειρά ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να κλείσουμε τώρα το θέμα, αλλά για δύο λεπτά έχετε το λόγο, κύριε Διευθυντά. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί γενικώ είναι πολύ θετική η στάση της ως προς την πρότασή μας. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με το δεξί. Και όσον αφορά το σύνολο του τοπίου υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο θέλω να σταθώ. Το ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι διεθνείς δεσμεύσεις και τα σχετικά με την επαναπρόθεση. Και στους τερμές διαλόγους λέγαμε τότε ότι θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα να προσθεθούν σε κάθε άρθρο της πρότασής του. Ε, βέβαια αυτό δεν συνέβη, αλλά έχουμε όλες τις ε, ρήτρες διαφύλαξης του ΣΥΠΗΝ σε σχέση με αυτό. Παρακαλώ, ρίχτε μια από τις προτάσεις μας. Δεν πειράξαμε καθόλου καθόλου αυτές τις ε, εξασφαλίσεις. Όχι, δεν κάνουμε πίσω γύρισμα σε αυτό. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. 100% σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για κάθε λειτουργία της υπηρεσίας και σε τρίτες χώρες. Αν θέλει περισσότερες ε, ρήτρες διαφύλαξης, ε, το κοινοβούλιο συμφωνούμε. Για την Τερμίλερ κάπως πιο επιφυλακτική στάση είχατε. σε σχέση με το ότι θέλουμε αυτήν την ε, πιο αναβαθμισμένη μορφή της συνοριοφυλακής και ακτοφυλακή. Ε, βέβαια, πιο το θέλει μια που μηχανισμός, οι ανθρωπινοί πόροι ε, στην πράξη δεν αποδίδουν. Το σύστημα δεν λειτουργεί. Άρα δεν μπορεί να αποδώσει όπως θα όφιλε η υπηρεσία. Απαράδεκτο. Και έχουμε εκπονήσει ένα σύστημα με τις τρεις κατηγορίες φαίνεται περίπλοκο, αλλά στι τεχνικέ αντίθεσει μπορούμε να σα εξηγήσουμε και την τελευταία λεπτομέρεια για το πώ αυτό το σύστημα θα παράσχει Το πώ θα έχει αυτέ τι 10.000 η υπηρεσία στη διάθεσή τη. Άρα αυτό χρειάζεται, χρειάζεται να τροποποιηθεί ο κανονισμός για το Eurosol και να γίνει σχετική αξιολόγηση γιατί για συνοριοφυλακή και εκτοφυλακή. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση που να έχει κάποια συνοχή για να λειτουργήσει, να είναι στεγανή ρύθμιση. Αυτό λέμε για νέο κανονισμό. Νέο, νέο κανονισμό. Αναβάπτεση <laughs> του κανονισμού. και για τις επιστροφές γιατί έτσι θα είχαμε τέτοια μορφή της πρότασής μας. Πρόταση 450 σελίδων της Επιτροπής. Με όλες τις μεταβολές. Αυτό θα είχαμε. Ε, αυτό όμως δεν θα μπορούσε να αποδώσει. Και γι' αυτό λέμε αντί της τροποποίησης να έχουμε καινούργια εκδοχή του κανισμού. Αντιγράφουμε τις υπάρχουσες διατάξεις. Δεν καθόμαστε να επανεφεύρουμε τον τροχό για κάθε επιμέρους ρύθμιση. Εδώ και δύο χρόνια αποφασίστηκαν αυτά από τον συνομοθέτη. Το θέμα της, επιτρο... της ε, της στην ε, επιστροφή. Ήταν από τα τελευταία θέματα που συζητήσαμε στον τριμερή διάλογο. Όπως έχει σήμερα η γεωπολιτική κατάσταση, θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Δεν λέμε ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει από την πρώτη στιγμή να πει ναι, αλλά οι συνομοθέτες αυτό το απέρριψαν πριν από δύο χρόνια. Ε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό δεν θα ξαναζητηθεί τώρα. Θα σας εξηγήσουμε γιατί ξανανοίγουμε την κουβέντα. Και θα δείτε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι ή αν δεν το δείτε θα πείτε όχι εμείς εμένουμε στα του 16 δεν θέλουμε να υπάρχει αυτού του είδους υποστήριξη επιστροφών. Αυτό θα σκέψουμε για το πόσο δηλαδή είναι βάσιμο να τροποποιηθεί ο βενζός. Α, είπονται κάποια άλλα ζητήματα και για το φάντο, ναι, με μεγάλη μου ευχαρίστηση να σας τα πω, αλλά μια που μου δώσατε δύο λεπτά, ε, τεχνικό είναι το θέμα, αλλά να τα πούμε, οι δυο μας. ή σε αυτές τις ε, τεχνικές συναντήσεις που τι επόμενες μέρες ή εβδομάδες πρόκειται να κάνουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ λίγο Πρόεδρος. Ε, Σκιώδη, είπαν ότι θα ξεκινήσουν αμέσω μετά από τη συζήτησή μα εδώ με την συνάντησή του. Περνάμε όμω εμεί στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή μα. Σημείο 3. Έκθεση της Eurojust για την χρηματοδότηση των τρομοκρατικών ενεργειών. Ο κύριος Λέναρτ, μέλος του Λουξεμβούργου στην Eurojust. So, you have 10 minutes, I think. Yeah? So,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 παρουσίαση της έκθεσης της Eurojust για τη χρηματοδότηση της δημοκρατικής ενέργειας. Παρόμοιες εκθέσεις εκδίδονται για υποθέσεις, την ομολογία, τη δικονομία μάλλον και τα σχετικά νομολογία. και τα σχετικά ένδικα μέσα. Ευχαριστούμε κύριε Λένα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. μου ζήτησε η ομάδα της Eurojust να σας παρουσιάσω τελευταία στοιχεία της έκθεσης αυτής για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τέλος πάντων δεν θα έλεγα ότι είναι και προσφατότατη, διότι είναι και εξημενών. Αλλά βασικός στόχος αυτής της πρότασης είναι να εξηγήσει τι κάνουμε για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό που δεν θα βρείτε εδώ είναι εξολόγηση κινδύνου. Οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Δεν είναι δουλειά μας. Πολύ θα ήθελαν ε, μερικές μυστικέ πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να τις δημοσιοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα συνεργασία. Πώς θα τους βοηθήσουμε να ερευνήσουν. Ό,τι άπτεται στι τρομοκρατίες βέβαια. Είναι μυστικού χαρακτήρα απόρριτου είναι πολλές οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, αστυνομικέ, διοικητικέ αρχέ, μυστικέ υπηρεσίες και το καθεξής. Δεν είναι κάτι το απλό. Εάν δει κανείς τις υποθέσεις αυτές καθεαυτές, βλέπουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν θα περάσω τώρα σε <coughs> αφηγήματα για το τι έχει συμβεί με την κάθε υπόθεση. Έχω επιλέξει κάποιε υποθέσει για να δείξω τι μπορούμε να κάνουμε. Η έκθεση απευθύνεται πιο πολύ στου συναδέλφου μα για να του πούμε ότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να έρθετε σε εμά. Έχουμε τώρα την σωρευμένη εμπειρία για να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επικεντρωνόμαστε στους ξένους μαχητές και την τάση αυτή και εκεί βλέπουμε υποθέσεις που έχουν σχέση με τρίτες χώρες, το δίκτυο των σημείων επαφής που βοηθά σε αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα, Δεν υπάρχει εγγύηση συνεργασία στον τομέα αυτό Απλώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι βοηθάμε τους συναδέλφους μας όσο πιο πολύ γίνεται. Επίσης στην έκθεση αυτή βλέπετε πώς βοηθάμε με τις διτακτικές επιστολές Λόγω της ε, σύστασής μας είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη από νομική σκοπιάς, αλλά και λόγω εμπειρίας. Και σε υποθέσεις που ανέφερα ε, ανέ, ε, και που αναφέρονται στο πρώτο τμήμα της έκθεσης, έχουμε καταφέρει να βοηθήσουμε. Να πούμε στους αδέλφους τι πρέπει να κάνουν για να προσάγουν κάποιους την δικαιοσύνη. Υπάρχουν μέρη του κόσμου που όλα αυτά είναι πιο περίπλοκα. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα πως σε μια ανθρωποκτονία ή κάτι τέτοιο. Αλλά ε, ασχολούμαστε με εγκλήματα ιδεχθεί όπως αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν και κοινέ ομάδε έρευνα, άλλο ένα ευαίσθητο θέμα στον τομέα αυτό. Μα χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να τελειοποιήσουμε τη συνεργασία με του συναδέλφου. Δυστυχώ, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στι Βρυξέλλε, α πούμε, έφτασαν πολλέ υποθέσει στα χέρια μα. τι ανέθεσαν πολύ γιατί μα εμπιστεύονται. Και έκτοτε έχουμε την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να βοηθήσουμε συναδέλφους εμπιστοσύνη διότι συγκεντρώνουμε πληροφορίες από πηγές που είναι μυστικές. Οπότε όταν συναντιούνται οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν με mail και γράμματα. Θέματα στρατηγικής, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμηθούν ε, κάποια φαινόμενα. Οι live, οι διαζώσεις συναντήσεις είναι οι καλύτερες. Δεν είμαστε ακόμα ένα στάδιο μεταξύ της συνάντησης κάποιων ξέρω εγώ, μια υπηρεσία στη Γερμανία και στην Αυστρία, τους βάζουμε στην ίδια αίθουσα να συζητήσουν για να δουν τι πρέπει να κάνουν. Η εγκύτητα με την Ευρωπόλ ήταν επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που αναπτύσσεται στην έκθεση. Ανέφερα τα τρίτα κράτη. Έχουμε συνεργασία και με τη ΣΥΠΑ, πολύ σημαντικό και αυτό το τομέα, ε, και άλλα σημεία επαφής και βοηθούμε και οικονομικά. Θα έλεγα ότι οι πόροι ε, λείπουν από τα κράτη-μέλη και όσο πιο πολύ συγκεντρώνει κανεί τι δυνάμεις του, τόσο πιο εύκολο μπορεί να καταπολεμήσει τέτοια φαινόμενα. Αυτό για το πρώτο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα θα τα δείτε. Υπάρχουν κάποιες υποθέσει, ως παραδείγματα. Και για να δούμε τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Από το ΠΚΚ μέχρι τον ΤΑΕΣ, το Άιζελ, όπως θέλετε πείτε το. Είδαμε πώς χρησιμοποιούνται τα αποδεικτικά στοιχεία. Τις διτακτικές επιστολές και πώς λειτουργούν, γιατί και αυτό είναι το κάτω δικαίου. Και μετά τη χρηματοδότηση που πρέπει να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ενέργεια ή όχι θα δείτε ότι τα ποσά είναι μικρά. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι 15.000. Δεν θα βρείτε εκατομμύρια να χρηματοδοτούν τις δράσεις. Αυτό βέβαια κάνει και την έρευνα πιο δύσκολη για τα κατημέλη. Και πάλι, ο στόχος του εγγράφου είναι να δώσει κάποιες παραμέτρους στους επαγγελματίε του κλάδου για να και για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα της εικόνας του τι συνολικά συμβαίνει. και δείχνει ότι έχουμε και τους πόρους και τις γνώσεις και τον τρόπο να εγγυηθούμε την εμπιστευτικότητα και τη μυστικότητα στον τομέα αυτό. Στο τελευταίο τμήμα θα βρείτε ένα μέρος της νομοθεσία μας. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο ενδιαφέρον τμήμα αυτό. Ήταν μια σύντομη παρατήρηση, παρά, παρουσίαση, συγγνώμη, αλλά αν έχετε ερωτήσει, είμαι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα. Υπάρχουν ερωτήσει από του συναδέλφου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Εάν όχι, Ήσασταν πολύ γρήγορο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ε, σημαντική δουλειά σα. Σίγουρα οι δραστηριότητες σας έχουν μεγάλη σημασία και αυτό φαίνεται και αν υπέθετε κανείς ότι δεν υπήρχατε τι θα γινόταν με αυτά τα θέματα. Αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να σα ευχαριστήσω. Thank So a... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν. Μέχρι τις 4.30, οπότε θα συνεχίσουμε το σημείο 4. Συνάδελφοι. να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένετε. Περιμέναμε προκειμένου να καταφτάσουν ο Σκιώδης και ο εισηγητής και και έτσι περνάμε στο σημείο 4 τη σημερινή διατάξη σε ό,τι αφορά του κανόνε με σκοπό τη διευκόλυνση τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, ανέγνευση, διεύρυνση, διερεύνηση συγγνώμη, ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αντικειμάτων. Και σήμερα έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, μάλλον όχι στον κύριο Ράδευ που είναι συγγετής, αλλά τον κύριο Λέραντς που τον αντικαθιστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και έχετε δίκιο. Έχω την τιμή να αντικαθιστώ τον κύριο Ράντεφ, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να προβληθεί σήμερα, αλλά θα διαβάσω την δήλωση που μου διαβίβασε σε διάφορε περιστάσει. Εμεί, ω μέλη του Κοινοβουλίου, βοηθήσαμε για την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για την καταπολέμηση σημαντικών εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία. Η έλλειψη α, τέτοιων πληροφοριών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ε, την ανικανότητα να, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τέτοιων εγκλημάτων και σε πολλές περιπτώσεις είμαστε σε αδιέξοδο γιατί δεν υπάρχουν εγκαίρως οι σωστέ πληροφορίες. Για να απαντήσουμε λοιπόν στις προκλήσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε άμεση πρόσβαση στα Μητρώα Εθνικών Πληροφοριών για τις αρμόδιες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της Europol και των εθνικών υπηρεσιών και αυτή η πρόταση διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ε, ΣΔΟΕ και των ε, μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών και της Europol σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή τέτοιων απόψεων και την ε, παροχή προθεσμιών για την απάντηση στα αιτήματα αυτά. Καλώ ορίζει λοιπόν ο εισήγητη την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρόκειται σε, για ένα βασικό ζήτημα για την καταπολέμηση ξεπλήματο χρήματο και άλλων σοβαρών ποινικών δοκιμάτων. Και καλώ ορίζει λοιπόν ο εισήγητη την διαταξή για την πρόσβαση στα εθνικά μετρώα και στα εθνικά μετρώα ανά πληροφοριών και των φορολογικών ε, συστημάτων, γιατί βασίζεται και στην πέμπτη οδηγία για τις ε, φοροαποφυγή και συμφωνεί η ανταλλαγή πληροφοριών ε, στην καταπολέμηση σημαντικών πενικών δικημάτων θα πρέπει να ενισχυθεί. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα συστήματα στα κράτη-μέλη και ότι πρέπει να διατηρηθεί η λειτουργικότητα και η αυτονομία και η ανεξαρτησία των αστυνικών σημάτων θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης από τις ε, αρμόδιες αρχές και από την Europol, λαμβάνοντα υπόψη κατά πόσο ε, μπορεί να υπάρχει και αρνητικό αντίκτυπος στις έρευνες από την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών ή κατά πόσον η κατα ποσο η αποκαλυψη των πληροφοριών αυτών είναι δυσανάλογη ή ενδεχομένω και άσχετη με το σκοπό για τον οποίο ζητείτε. Προθεσμίες ε, για την χορήγηση πληροφοριών έχουν παραταθεί κατά της για να υπάρχει ένα περιθώριο δράσης και τέλος ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων υφίσταται ήδη και θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία νέων τέτοιων πλαισίων. Ο κ. Ράντεφ επίσης ήθελε να δηλώσει ότι οτιδήποτε σχόλια εκφράσουν οι συνάδελφοι θα του διαβιβαστούν και ότι προσβλέπει φυσικά στη συνεργασία με τους συναδέλφους στο θέμα αυτό και ότι η προθεσμία έχει, για την κράτηση τροπολογιών έχει, έχει οριστεί η 19η Οκτωβρίου. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, εξ ονόματος της ε, Κατερίνα Τσινίτσι, η κυρία μυρια μνταλη το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς εξ ονόματος της κυρίας Κινίτσι θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της ε, για το γεγονός ότι απουσιάζει είχε προανειλημμένες θεσμικές ε, υποχρεώσει στην Ιταλία. Ευχαριστεί τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση που παρουσίασε. Εκφράζει εκτίμηση για τις ιδέες που υποβληθήκαν στο κείμενο όπως και πιο πολλοί συνάδελφοι, συμφωνεί με τους στόχους ε, της πρότασης και το στόχο διευκόλυνσης μιας ε, καλύτερης ανταλλαγής και πιο ευκολότερης ανταλλαγής ε, πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των εθνικών κρατών μελών και της Europol, δεδομένου μάλιστα και του διεθνητικού διεθνικού χαρακτήρα των εγκλημάτων αυτών θα πρέπει να υπάρχει έγκυρη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων για άτομα τα οποία υποπτευόμαστε ότι έχουν διαπράξει σοβαρά δικαίωματα τι επόμενε εβδομάδες. Η κυρία Κινίτσι θα αναζητήσει σωστή ισορροπία μεταξύ των ισορροπιών και των αρμοδιοτήτων της κάθε υπηρεσία, προκειμένου να υπάρχει πιο αποτελεσματική δίωξη τέτοιων αδικημάτων. Η κυρία Κινίτσι στο πλαίσιο αυτό εκτιμά το γεγονός ότι έχει εισαγάγει ο εισηγητής ε, κάποιες ε, ε, διατάξεις λοιπόν, για την προστασία των εθνικών αρμόδιων αρχών και θέλει να δοθούν εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προτείνεται και από τον ε, σχετικό Ευρωπαίο επόπτη και πιστεύει ότι είναι κρίσιμη σημασία να υπάρχει σωστή εκπαίδευση των ατόμων του προσωπικού που έχουν στα χέρια τους τέτοια προσωπικά δεδομένα και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τη διαδικασία ε, ε, της πληροφοριών σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με την Europol και πιστεύει ότι οι, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ακολουθήσουν ε, τις ε, προδιαγραφές της πέμπτης οδηγίας για το ψέπλωμα χρήματα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία τους και πιστεύει παρ' αυτά ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία τους και η κυρία Κνήση πιστεύει ότι ο στόχος ε, για οι στόχοι μάλλον που θα πρέπει να καλύπτουν τα θέματα για τα οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίε πρέπει να οριστούν. Και επίση να ληφθεί υπόψη πώ δεν θα διακυβεύονται οι τρέχουσε έρευνε και στα πλαίσια τη συνεργασία με τη Πόλη είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε σωστό συντονισμό με τι εθνικέ αρχέ, που είναι υπεύθυνε για την δημόσια ασφάλεια προκειμένου να κοινοποιούνται τέτοια αιτήματα για πληροφορίε. Κύριε Κινίτσι πιστεύει ότι η προθεσμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ανταποκριθούν οι εθνικέ ε, υπηρεσίε, θα πρέπει να ε, παραταθούν, να διευρυνθούν για να μην δημιουργηθεί αρνητικός αντίκτυπος και να μην υπάρχει και αρνητικό αντίκτυπος και στην ποιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται τέλος. Θα πρέπει να σκεφτούμε τον ορισμό των εγκλημάτων για τα οποία μπορεί να ζητήσει η Europol ε, τη χορήγηση τέτοιων πληροφοριών από τις Εθνικές Αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Μυρία λέει ο Πρόεδρος. Η Έλκα Στίβενς τώρα είναι η επόμενη σκιώδη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλησπέρα στους συναδέλφους. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης, για το σημαντικό αυτό θέμα. Και θα ήθελα αυτής εξ αρχής να πω ότι η έκθεση αυτή είναι ισορροπημένη και αναγνωρίζει ε, πώς έχει η κατάσταση στα εθνικά κρατή-μέλη σήμερα, οι εγκληματικέ Οργανώσει. Ε, έχουν ε, τις δράσεις τους και τους λογαριασμούς τους ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία για να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ διαφόρων ε, λογαριασμών και νομισμάτων με πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού. Στην καταπολέμηση λοιπόν κατά του οικονομικού εγκλήματο, οι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι απαραίτητο ο ρόλο του να μην ε, αλλάχθει παρά μόνο όπου είναι αυτό απολύτω απαραίτητο. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επηρεάσουμε την ανεξαρτησία και την αυτονομία των ε, μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ελεύθερα τις δράσεις τους και αυτό συμπεριλαμβάνει τη λήψη αυτόνομων ανεξάρτητων αποφάσεων για τη διαβίβαση μη πληροφοριών. Πέραν τούτου, πιστεύω ότι η υποχρέωση για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών συμβάλλει στην ε, πιο γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση τέτοιων δοκιμάτων. Και τέλος, αναγνωρίζω ότι είναι σχέση μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και της Europol, αλλά έχω αμφιβολίε για το πόσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η δέσμευση για τι μονάδες τις εθνικές αυτές μονάδες. Όπως βλέπετε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε ακόμα και προσβλέπω σε αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η πρόταση, γιατί είναι στο μικρό των δικών μα προτεραιοτήτων όσον αφορά καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματο και τη τρομοκρατία. Αυτή η πρόταση βελτιώνει την ανταλλαγή των πληροφοριών μόνο σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη γίνεται ε, ανταλλαγή πληροφοριών από το δίκτυο αυτών των πληροφοριών που το διαχειριστεί η Νομίζω ότι είναι τώρα μια ευκαιρία με αυτή την οδηγία να έχουμε ε, κάποιο είδους τέτοια ε, μονάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να λειτουργεί ετής ενδιαφερόμενο και έτσι να μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα πιο φιλόδοξο, να έχουμε επομένω περισσότερους πόρους και καλύτερο συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιμέρους τέτοιων μονάδων. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να ελαμβάνει τα μηνύματα για τις επιλήψιμες συναλλαγές η Ευρωπαϊκή Μονάδα, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά είναι θέμα ελεγού και συντονισμού. Επίσης είναι και ζήτημα προστασίας των δεδομένων που αναδύεται εδώ, γιατί έχουμε μια σειρά άρθρων που εγκρίνουν κατά κάποιο τρόπο την επεξεργασία κάποιων δεδομένων, προσθεντολισμό και λοιπά. Όλα αυτά μπορεί να τα επικαλείται κανείς σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν χρειάζεται εδώ νόμος ειδικό ο οποίος να αποκλίνει από τον γενικό κανονισμό ε, για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε την οδηγία 680 ε, του 16 που ήδη ορίζει ε, ποιε είναι οι εξασφαλίσει όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα και οπότε θα πρέπει η πρόταση εκεί να παραπέμπει. Επίσης με πάρα πολύ θετική την στροφή που γίνεται από το εισηγητή την έκθεση. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνονται οι απαντήσεις ε, στις αιτήσεις υπαρχής πληροφοριών. Θα πρέπει να είναι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών η ταχύτερη δυνατή μεταξύ των αρμοδίων μονάδων και των αρμοδίων άλλων αρχών και δεν θα πρέπει ε, να, να μπαίνουν τροχοπέδι καθυστερήσεις στη δουλειά των ε, μονάδων αυτών. Δεν θέλουμε να φύγεται η ανεξαρτησία και η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση σε περίπτωση άνθρωσης παροχής πληροφοριών. Πάντως θα πρέπει όλες οι επιλογές να εξετάζονται με προσοχή. Ας συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με αυτή την πρόταση για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση όσον αφορά την καταπολέμηση αυτών των ε, εγκλημάτων και γενικότερα την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο Ζεράρ Ντεπρέ για την Άλντε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την απουσία του σκιώδους μας, κύριο Πέτρισεν ο οποίος δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Συγγνώμη εκ μέρους του. Ευχαριστά, ευχαριστεί τον εισηγητή για τη δουλειά του. Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονό ότι το θέμα της διαφοράς το μεταξύ των επιτροπών έχει επιληθεί για να γίνει σωστή δουλειά για την έκθεση αυτή από τώρα. Ε, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών για την καταπολέμηση αυτού του είδου εγκληματικότητα και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών με τον πλήρη σεβασμό όμω των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ο Σκιώδης μας εκφράζει μια ευχή. Επειδή είναι πολύ σύντομη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και πρέπει να εργαστούμε βιαστικά, να μας δοθεί λίγος χρόνος παραπάνω. Με αυτά σας έχω μεταφέρει το μήνυμα του εισηγητή μας. Ευχαριστούμε. Κοιτάζω αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει ακόμα το λόγο. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος να σχολιάσει. Η Επιτροπή, παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Είμαι ούτε Στεγκέλ, υποδιευθύντρια από την DG Home. Τα έχουμε εξετάσει και με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Τρανς. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που έχετε προωθήσει αυτό το θέμα. Την πρόταση την υποβάλαμε φέτος τον Απρίλιο με σκοπό έγκριση να έχουμε πριν τις ευρωεκλογέ του χρόνου. Νομίζω μπορούμε να έχουμε την ε, πεποίθηση ότι αυτό θα συμβεί. Με βάση το πρόγραμμά σας. Από την πλευρά μου να πω ότι είμαι χαρούμενη Χαίρομαι που ε, σας αρέσει η άμεση πρόσβαση για τις διοκτικές αρχές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Και χαίρομαι πολύ που δεν υπάρχουν τροπολογίες για τις διατάξεις αυτές. like Να πω και εγώ δύο λόγια το όνομά μου είναι Δέσποινα Βασιλιάδου. Είμαι υποτινατάρχη στην καταπολέμηση του οικονομικού κλίματος στην ε, Γενική Διεύθυνση Τσάστ. Άκουσα πολλά σχόλια σήμερα για το θέμα. Να πω ότι η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών ε, οικονομικών πληροφοριών, δίωξη οικονομικού εγκλήματο δηλαδή και διεκτικών αρχών. Στόχο τη πρόταση που βάλαμε είναι να ενισχύσει τη συνεργασία. Και άκουσα από όλου στην αίθουσα ότι σα αρέσει και ότι θέλετε ενδυνάμωση τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών δίωξη οικονομικού εγκλήματο και διοκτικών αρχών. Παρ' όλα αυτά, αν δω το σχέδιο έκθεση πρέπει να παραδεχτώ ότι ανησυχώ λίγο. Οι υποχρεώσει ε, συνεργασίας διαγράφησαν και αντικαταστάθηκαν από μια ρήτρα που επιτρέπει την ανταλλαγή. Οι ανταλλαγέ επιτρέπονται και σήμερα με την τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Ανησυχώ λοιπόν κάπω ότι με τι τροπολογίε που έχουμε μπροστά μα σήμερα Τελικά δεν ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ακριβώς την ίδια μορφή συνεργασίας που ισχύει και σήμερα. Πολλοί αναφέρεται την ανάγκη να έχουμε ανεξάρτητες και αυτόνομες αρχές ε, οικονομικού εγκλήματος Αλλά θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολιτική ανεξαρτησία, να μην υπάρχουν παρεμβάσεις. και ανεξαρτησία αυτονομία, αλλά όχι άρνηση ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες κυβερνητικέ αρχές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν είναι αυτό ανεξαρτησία για μας. Επίσης να πω ότι όταν υποβάλαμε αυτή την πρόταση θεωρούσαμε ότι απαντούμε σε αιτήματα του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αρχών δίωξης οικονομικού εγκλήματος και διοικητικών αρχών. Αυτό το αίτημα μας φάνηκε να το έχουμε ακούσει και βάσει της έκθεσης της Επιτροπής για το σκάνδαλο Panama Papers και τα σχετικά πορίσματα. Και υπήρξε και άλλη μια έκθεση που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτο για την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία που ζητά κάτι παρόμοιο. Η διάσκεψη των Παρισίων από φέτο το Απρίλιο ε, ζητούσε επίση κάτι ανάλογο, περισσότερη συνεργασία μεταξύ των FIU και των διοικητικών αρχών. Αυτό λοιπόν θεωρούσαμε ότι κάνουμε. Χάρη που άκουσα ότι δεσμεύεστε πολιτικός για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα και να αντικατοπτρίζονται και στην νομοθεσία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών, με κάποιε εξαιρέσει βεβαίω που μπορούμε να τι συζητήσουμε, αλλά η υποχρέωση συνεργασία πρέπει να είναι δεσμευτική, όχι απλώ να δίνεται μια δυνατότητα. Ανυπομονούμε να δούμε τι τροπολογίε των σχεδόν εισηγητών σα και να συνεχίσουμε τη συνεργασία, μα. συνεργασία μα. Ευχαριστώ πολύ που μα δώσατε το λόγο. So Ωραία. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Να πω αυτό που μας είπε και ο εισηγητής. Δεδομένης της σημασίας του θέματος πρέπει να επιταχύνουμε για να προλάβουμε να το ολοκληρώσουμε πριν την ε, λήξη της θητείας. Αυτό είναι το πλαίσιο του οποίου ο εισηγητής προτείνει μια διαφορετική διαδικασία. Και μάλιστα η προθεσμία πρέπει να αλλάξει από τις 19 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα που προβλέπετε τώρα. Αυτό θα σας πω ότι ούτως ή άλλως μόνο ο συγκεκριτής μπορεί να το αποφασίσει. Προθεσμία επισήμως λοιπόν 19 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Το ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο και πάλι έχουμε ελεύθερο χρόνο. Ο πρόεδρος είναι κάπου εδώ στο κτίριο και θα έρθει για την ψηφοφορία.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 Uh, dear colleagues, um, we'll be voting at 17.15. Πέντε και τέταρτο συνάδελφοι θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Σιγουρευτείτε οι αναπληρωτές ότι έχουν τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Συνάδελφοι που δεν ψηφίζουν συνήθως δηλαδή. Συνοηθείτε με το επιτελείο σας να βεβαιωθείτε ότι έχετε την κάρτα. 5 και 4, άρα να είστε όλοι. Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, λείπουν, λείπουν συνάδελφοι από περισσότερες ομοιοπολιτικές ομάδες. Είναι σημαντικό, οπότε και θα πρέπει να περιμένω. Λείπουν πάνω από μιας ομάδας συνάδελφοι. Άρα η υπομονή για ολίγων λεπτών. Κορνίλια, do you have a point of order? έχεις διαδικαστικό, κυρία Έρνστ. Δεν έχω την κάρτα μου, λέει η κυρία Έρνστ. Α, τη χρειαζόμαστε. Μήπως μπορεί κάποιος να πάει να στη φέρει από τον τρίτο. Κάποιος από την ΚΟΥΕ, παρακαλώ, ας φέρει την κάρτα της κυρίας Έρνστ. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε να έρθουν συνάδελφοι. Τι χρειαζόμαστε. Can I just, um, colleagues, just let me make a check, please, that everyone who is present has their electronic voting card. Σιγουρευτείτε ότι την έχετε, συνάδελφοι όλοι που είσαστε εδώ και πρέπει να ψηφίσετε. Ιδίω οι αναπληρωτέ. Μόνο η κυρία Έντζ δεν έχει. Καλά, θα, θα τη φέρουν. Δεν θέλω να αρχίσουμε να υπολογίζουμε ψήφους Χωρί κάρτα. Από τον τρίτο, ε. Στον τρίτο δεν είναι. Κάποιος θα πάει να στη φέρει. We'll make an arrangement if we can't get it on time. Καλά, θα τα βρούμε αν δεν μπορέσει να έρθει γύρω. Έρνστ. Δεν την έχω, αλλά ο συνάδελφος θα πάει να τη φέρει εδώ. Αλλά θα σας ε, κάνω νόημα για το τι ψηφίζω. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι Κονιλία. Θα στη, θα στη φέρουν και αν αρχίσουμε θα σημειώνουμε το τι ψηφίσεις. Αν βέβαια οι συνάδελφοι δεν έχουν αντίρρηση. Δεν ξέρω τώρα να δούμε. Να ε, σιγουρευτούμε ότι δεν είναι άλλο στην ίδια κατάσταση μέσα. Ωραία. Συνάδελφοι. Λείπουν, λείπουν συνάδελφοι από περισσότερες πολιτικές ομάδες. Έρχονται. Είναι καθοδόν. Γι' αυτό αν συμφωνείτε να τους περιμένουμε. Yes.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 um, can I speak to someone from the e group? Για να μου πει κάποιος από την Γκουέ. Ε, e. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε για να μην στρεβλώσουμε την ψηφορία. Για κοιτάξτε. Λείπει κι αλλουνού η κάρτα. Λείπει. Έρχεται η κάρτα. Έρχεται. Δεν θα αναφέρω κανείς σε δυσκολίε, αλλά θα είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία μα εφτάκτω. Οι συντονιστέ τι λένε, είναι εδώ, ωραία. ΕΛΚ, Άλντε. Um, Ποιο είναι σήμερα, Σόφια. Εσύ αντικαταστάς τον συντονιστή. Εντάξει είσαστε στην Άλντε. Όλοι εδώ. Okay, I take it that genial chuckle that everything is fine. Α, βλέπω από τα γελάκια σας καταλαβαίνω ότι όλα καλά. Γκουε, πράσινη, όλα καλά, ECR. No problem. Χέλγα.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 I'll make an announcement for the one voting card that is not here, and I'm sure it's on the way uh, before we start voting. Θα έρθει η κάρτα πριν αρχίσει η ψηφορία. Εγώ κάνω τις ανακοινώσεις μου στο μεταξύ. Thank you, colleagues, for... Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Οπότε μιλάμε τώρα για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφόρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύνορα και θεωρήσει. Έχουμε συνεισηγητέ, Λέναρ και Μέλο. Θέλουν οι εισηγητέ τον λόγο πριν αρχίσουμε να ψηφίσουμε. Όχι. Ωραία. Οπότε πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε στην πρώτη στήλη και θα σας λέω, θα σας διαβάζω μάλλον. Της τροπολογίας. 195 ψηφίζουν. Okay, colleagues, so the EPP has two plus. So if... Δύο παραπάνω στο ΕΛΚ. Δύο πρέπει να αποσυρθούν για να κάνουμε την καταμέτρηση. Ναι, οκ, ωραία, ωραία, τώρα είναι εντάξει. Closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεν ξεκινήσαμε με το δεξί, βλέπω. 196, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 197 ψηφίζουμε. Εντάξει είναι, το, το πάω αργά αργά. Ψηφίζουμε ακόμη. Um, as everyone voted, the vote is closed and that's rejected. Απορρίπτεται. Mm. Κάποιος σηκώθηκε και έφυγε. Έφυγε κάποιος νηστής. Πω πω. Είπατε ότι είμαστε δύο παραπάνω. Φύγανε τρεις, άρα λείπει ένας. Τρία πλην δύο, α, να, να, να, ξαναγύρισα. Θέλετε να περιμένουμε μέχρι ότου να επιστρέψει ο συνάδελφος που έφυγε. Ε, δεν ωφελεί κανέναν. Α, ήρθε, ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα α συμβαστική. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Πέρας. Εγκρίνεται. 386. Ψηφίζουμε. 386 στην πρώτη στήλη. Σελίδα 5. Πρώτη σελίδα 386. Ψήφισαν όλοι. Πέρασαν. Εγκρίνεται. Άρθρο 3. Και τροπολογία 391. Δεύτερη στήλη. 391 ψηφίζουμε. 391, το ακούσατε όλοι. Στο 6, άρθρο 3. Επαναλαμβάνω. Άρθρο 3. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Δεν τελειώσαμε. 391. Ernst. Το ότι όλοι πέρας Παρακάτω, 399. Πάντα είμαστε στο άρθρο 3. Απαλληφή. Έρνστ. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 400. Νίτερ Μιλερ. Ψήφιζαν όλοι Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική Τρία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Συμβιβαστική. Τέσσερα. Ψήφιζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τετρακόσια εννέα. Ψηφίζουμε. Τετρακόσια είκοσι εννέα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πέντε ψηφίζουμε. Εγκρίνεται συμβαστική 6. Πέρας. εγκρίνεται 443 πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 7 ψηφίζουμε Vote is closed. And that's carried. Compromise Amendment 8. Vote is open. 8. Ψηφίζουμε.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 Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 535. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 539. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι. Α, στο 73 λέει γραμματέας. 73 ψηφίζουμε. Εβδομήντα του άρθρου 19, στη σελίδα 20. Το ακούσατε όλοι, 73. Πέρασε. κρίνεται. Δέκα επτά. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται 569 σελίδα 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. 18. Ψηφίζουμε. Συμβαστική 18. Ψηφίζουμε πέρας. Εγκρίνεται. 585 ψηφίζουμε. Vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Ψηφίζουμε. Τη σελίδα 29. Εκεί βρίσκεται η τροπολογία 21. Ψηφίσαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 609 ψηφίζουν. Επίσης τη σελίδα 29. Το 609. Πέρασε. Εγκρίνεται. Θα σας λέω τις ε, σελίδες γιατί αυτές είναι κοντά στο κείμενο. Όχι, όχι, έκανε λάθος. Δεν θα πρέπει να σας λέω τη σελίδα γιατί μπερδεύετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ψήφισα 613. Ψηφίζουμε. Όλες μαζί. Αυτές υπό το 613. Πέρασε. Εγκρίνονται. σημείο. 602, 614. 614-602 ταυτόσημες. το Ψηφίζουμε, περα Εγκρίνονται. Συμβαστική 22. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 622 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 622 επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Έτσι μου είπαν ότι το ψηφίζουμε. Ναι, ναι, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ταυτόσημες. Α, όχι. Λέει ο πρόεδρος. Και πάμε... 634. 634. λέει. Vote is closed. Πέρας.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 That's carried. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 ψηφίζουμε. Vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται συμβαστική 25. Ψηφίζουμε. Vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Ψηφίζουν. Πέρασε. Εγκρίνεται. 27. Ψηφίζουν. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ή 34. Άρθρο 34. Πάμε στην τροπολογία 110 του άρθρου 34. 110. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Ψηφίζουμε. Sorry, compromise amendment. Α, συμπαθάτε με γιατί παρέλειψε το 28. 28 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται συμβαστική 29. Πέρασε. Εγκρίνεται 30. Πέρασε. Εγκρίνεται. 702. Ψηφίζουμε. 702. Πέρας. Εγκρίνεται. 120. Εγκρίνεται. 31 ψηφίζουν. Εγκρίνεται 32. Ψηφίζουν. Εγκρίνεται το 615. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Στα Συγγνώμη, συνάδελφοι, πρώτα ψηφίζουμε τη συμβαστική 33. Ψηφίζουμε. Και κάποιες ταυτόσημες πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 41. Το 726, 727. Ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Κατόν τριάντα ένα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται συμβαστική 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 36. Υπέρ. Ε, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 45. 145. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 743. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 37 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Επτά, πέντε, οκτώ. πενήντα οκτώ, συνάδελφοι το ξέχασα, έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 40. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 41. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Άρχεται. Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβαστική 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. αγκρινεται 8. 2, 0, 820. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47. Υπέρ. Συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 175. 175. Unblock. Ομαδικά. έρχεται άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται. Άρθρο 55. 176 συνάδελφοι 176 άρθρο 55α, 176, άρχεται η ψηφοφορία. Άρθρο 55α. Εκατόν εβδομήντα έξι άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Γκρίνεται. 55 D. 178. Στη δική μου την ε, αρρύθμιση είναι σελίδα 60. Εσείς μπορείτε να το έχετε αλλού. 178 του άρθρου 55D. Το βρήκατε όλοι. Πέρας. Με συγχωρείτε, άρχεται η ψηφοφορία πρώτα. Τώρα πέρας. Εγκρίνεται. 179. 179. πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 40α. Άρχεται. Συγγνώμη, 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εννέα, τέσσερα, τρία, 943 περιμένω να 943 περιμένω να το βρείτε όλοι εμένα είναι 74 το δικό σας 79 943 στο άρθρο 56 της κυρίας Ιεντβέλτ. 74 έχω εγώ μπροστά μου, εσείς μπορεί να έχετε 79, λέει ο πρόεδρος. Το βρήκατε, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 49. Άρχεται η ψηφοφορία.

Εγκρίνεται. Και τώρα θα πάω αργά, γιατί είναι όλε. παρόμοιε. Άρθρο 58. Άρθρο 57, 958, του κυρίου Νταλτών. Πέρας. Απορρίπτεται. 58. 959, 960 ταυτόσιμες άρχεται. Μποντίλ Βαλέρο και Κορνίλια Έρνστ. Πέρας. Απορρίπτονται. Εξήντα προϋπολογισμούς. Όχι, με συγχωρείτε. Έχασα ολόκληρη συμβαστική. Συμβαστική, μετά από τόση σκληρή δουλειά. Συμβαστική 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Η 961 καταπίπτει εφόσον εγκρίθηκε η 959. Έτσι δεν είναι. Ξέρω ότι δεν πιστεύετε ότι έχω δίκιο, αλλά αλήθεια είναι. 50 λοιπόν, ακόμα ψηφίζουμε ενώ το ψάχνουμε. 50. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα. Όπως λέγαμε, τροπολογίες της Επιτροπής Προπολογισμών. Budget 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάτι έπαθε το μηχάνημα. Το μηχάνημα τα τίναξε. Είναι εξαντλημένο. Εγκρίθηκε αλλά δεν λέει τίποτα η δική μου οθόνη. Budget 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 3. Budget 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 973. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 981. Άου και Ζήλστρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 986 65 της κυρίας Ένστ. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 52. Συμβαστική 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 189 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 989. 989. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεστική 53. Άρχεται. πέρα. Εγκρίνεται. Budget 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Budget 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 199. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 200. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 201. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 202. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 206 άρχεται. Διακόσια έξι. Άρχεται η ψηφοφορία. Διακόσια στην άλλη στήλη, συγγνώμη, και του κυρίου Μέλου. Τώρα που το βρήκατε, ας κάνουμε αυτό και βλέπουμε. 206 του κυρίου Μέλου. 206. Στη στήλη του κυρίου Μέλου. Άρχεται. Πέρας. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 207 Ζήλστρα. Τα ονόματα τα λέω για να έχετε πιο πολύ χρόνο να ψηφίσετε, έτσι. Δεν για κανένα λόγο. Πέρας. Απορρίπτεται. 211 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. «210» στην κολόνα στη στήλη του κυρίου Μέλου. Έχει γίνει μπέρδεμα τώρα. Πέρας, απορρίπτεται. 214 άρχεται. Στη στήλη του κυρίου Λέναρς. Πέρας. Εγκρίνεται. 215. Πέρας. Απορρίπτεται. Διακόσια είκοσι εννέα. 229 Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 230. 230. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 232. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 236. Άρχεται. ...236... ...πέρας... ...απορρίπτεται... 249 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 276 τώρα άρχεται. Το βρήκατε όλοι 276. Ναι, ναι, το αφήνω. 276. Ωραία, ψήφισαν άπαντες, πέρα Απορρίπτεται. Τώρα 200... 290. 290. Για, τα, για το αρχείο μας είχα δίκιο πάλι, καλά είχα πει 289, 289, 289 πρώτα, 289, πέρας, απορρίπτεται. 290 άρχεται. 290, την ψηφίζουμε, πέρας. Εγκρίνεται, 291, έρχεται η ψηφοφορία. Καταπίπτει. 295, 295 τώρα. Πέρας απορρίπτεται. 296 άρχεται. Πέρας απορρίπτεται. 307. 307. Σα ευχαριστώ αν ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Η 10 παρακαλώ. Η 10, τροπολογία 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 3, 14, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 315. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Η 320 παρακαλώ. Η 320 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 321 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 322 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 12 παρακαλώ. Όχι. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Η 327. 327 ψηφίζουμε, παρακαλώ. Η 327. Ψηφίσατε, παρακαλώ, όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 328. 328 ψηφίζουμε. Α, μου ξέφυγε η 324, αλλά μόλις ολοκληρώσαμε την 328. Όχι, να ψηφίσουμε την 328, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την ψηφοφορία και μετά θα σας πω τι λάθος έγινε. Πέρας για την 328 εγκρίνεται. Και συνάδελφοι να πάμε πίσω στην 324, στην κυρία, στην τροπολογία Ντεπρέ, η οποία δεν εξαρτάται από τίποτε άλλο. Να ψηφίσουμε παρακαλώ το 324 που μας ξέφυγε. 324. Ζητώ συγγνώμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 14 λοιπόν τώρα. Η 14 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 335 ψηφίζουμε. 335. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Σας ζητώ συγγνώμη, η 334. 3-3-0-4 3.34 ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 3.34. Περάς. Απορρίπτεται. 335. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Περάς. Απορρίπτεται. Η 338 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 339. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 340. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και αυτή εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες. Η 3-2 και 345. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 347. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 348. Ψηφίζουμε. πέρας εγκρίνεται. Η 349 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 350 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 351. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα με ονομαστική κλίση παρακαλώ η τελική ψηφοφορία. Καταρχάς, έτσι τη λογικότητα για τα σύνορα και τη βίζα για τον κύριο Λέναρ. Έκθεση Λέναρ. Ε, ψηφίζουμε. Με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. πέρασα. Εγκρίνεται. 44 ψήφοι, 10 κατά, 45 μάλλον υπέρ, 10 κατά, 0 αποχές. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόφαση για την έναξη των διαπραγματεύσεων. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 43 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 2 αποχές. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο θέμα, τη διαλειτουργικότητα για την αστυνομική και αντικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση. Ο κύριος Μέλο, εισηγητής, ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, καμία αποχή. Και τώρα για την έναξη των διαπραγματεύσεων ψηφίζουμε, παρακαλώ. Έναρξη. Και πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και έτσι ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία και τη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ.